λόγο, με λόγια αλήθειας. Ότι σε όλες αυτές τις συνέπειες, τις αμέτρητες συνέπειες ε, του Brexit, σε όλους ε, τους τομείς, εγώ σας μίλησα με λόγια αλήθειας λοιπόν και γνωρίζουμε ότι μεταξύ όλων των αιτιών του Brexit ε, μία από τις αιτίε και ένα από τα κίνητρα των ίδιων των υπερασπιστών του Brexit. Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι. Ένα, ανάκτηση της δυνατότητας να αποκλίνουν και να παρεκκλίνουν ε, των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, φορολογικών ε, διατάξεων που ε, βρίσκονται στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και δεύτερος λόγος που μας επισήμεναν προηγουμένως είναι η... ο δραματισμός της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών που βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν την οποία αντιμετωπίζουμε και έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον. Όπως είπατε πολύ και θα το συζητήσουμε βέβαια και στις μελλοντικές διαπραγματεύσει θα υπάρξουν και συγκεκριμένες πολύ απτές συνέπειες σε ό,τι αφορά την ε, κατάργηση μετά την μεταβατική περίοδο, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα συγκεκριμένα καθεστώτα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά προσόντα, τη δυνατότητα εγκατάστασης και την ασφάλεια. Κανείς από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να υποτιμήσει, και από τις δύο πλευρές, έτσι, το επισημαίνω, δεν μπορεί λοιπόν να ε, υποτιμήσει τις άμεσες συνέπειες της κατάργησης αυτής της ελευθερίας ε, μετακίνησης που βρίσκεται στο επίκεντρο του Brexit. Αυτά σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ διαπραγματεύσει που θα ξεκινήσουν στις αρχές Μαρτίου. Προς το παρόν, μιλούμε για τα δικαιώματα των πολιτών, που είναι προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, αλλά και του Ευρωπαίου διαπραγματευτή. Σας ευχαριστώ. Αποτέλεσε επίσης προτεραιότητα όλων των κρατών μελών ε, τα οποία εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ τον κύριο Βερχόφστατ και όλους τους συναδέλφους για αυτό το εξαιρετικά σαφές ε, ψήφισμα που έχετε καταθέσει και εκφράζει ακριβώς ε, την επαγρύπνησή σας και την αλληλεγγύη σας προς τους πολίτες που πλήττονται από τις άμεσες συνέπειες του Brexit ο κύριος Βερχόφστατ ε, θα μπορέσει να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει, για να βασιστεί πάνω σε αυτή την ισχυρή πλειοψηφία για τις πραγματές που θα πάρουν ε, χώρα τι επόμενες ημέρες. Οι πολίτες, λοιπόν, όπως υπόθηκε, χρειάζονται βεβαιότητα, σαφήνεια για το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους. Θέλουν να ξέρουν τι ακριβώς θα σημάνει το Brexit για εκείνους και την καθημερινότητά τους. Αντικειμενικά, θεωρώ ότι η συμφωνία αποχώρησης που έχετε μπροστά σας παρέχει αυτή τη βεβαιότητα για τους ε, Βρετανούς ε, πολίτες ε, που διαμένουν σε ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρώσει πριν το τέλος της μεταβατικής περίοδου, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2020. Και έτσι θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πριν, στη χώρα διαμονής τους. Αυτό ισχύει για περίπου 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετέχουν στην ε, οικονομία και στην ανάπτυξη της ε, Βρετανική οικονομία. Όλοι αυτοί λοιπόν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται, να σπουδάζουν, να συμβάλλουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, να δημιουργούν ε, και να ζουν μαζί με την οικογένειά τους, να συνεχίσουν τι ζωές τους. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα αυτή τη ε, συνθήκης γιατί για συνθήκη πρόκειται με όλες τις νομικές ε, προεκτάσεις μετά την κύρωσή της και από τις δύο πλευρές. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να επακρυπνήσουμε για την σωστή υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Δεν θα δεχθούμε ημίμετρα και διακρίσεις, ακόμα και αν αυτές είναι συγκαλυμμένες. Είναι ευθύνη δική μου και της ομάδας μου ε, να επαγρυπνήσουμε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σωστή υλοποίηση αυτής της ε, συμφωνίας και μετά τη μεταβατική περίοδο φυσικά θα έρχομαι όσο συχνά θέλετε για να σας ενημερώνω για την ε, σωστή υλοποίηση ε, της συμφωνίας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις ε, ελευθερίες και τα συμφέροντα των πολιτών μας. Ευχαριστώ και τις 27 πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λονδίνο που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πολιτών μας και θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε την ε, πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας αποχώρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το παν για να διασφαλίσει τα δικαιώματα ε, του ενός εκατομμυρίου Βρετανών πολιτών που μένουν στα 27 κράτη-μέλη Θέλουμε να διατηρηθούν αυτά τα δικαιώματα, θέλουμε ε, όλοι τους να ενημερώνονται και να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη και θα εργαστούμε σκληρά ούτως ώστε και η Βρετανική κυβέρνηση να κάνει ακριβώς το ίδιο και για τα 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που μένουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήδη έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα σε ό,τι φορά το καθεστώ ε, εγκατάσταση ε, τη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν γύρει πολλέ οργανώσει πολιτών, αλλά σήμερα το αθήξατε και πολλοί από εσά. Καθώ και η υπόθεση της ε, Εμμανουέλ που ανέφερε η Καρολάιν Βόρντεν προηγουμένως. Η Επιτροπή με μεγάλη προσοχή θα παρακολουθεί ε, τι ε, υποθέσει συγκεκριμένων πολιτών και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν για την κατοχήρωση του δικαιώματο παραμονή του. Ε, φυσικά θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι πολίτες να ακολουθήσουν τις διοικητικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Βρετανική πλευρά. Έχουμε θίξει μία σειρά τέτοιων ε, προβληματισμών με τον ε, Στίβεν ε, Μπάρκλεϊ και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε, ιδίως ότι αφορά τη σημασία της θέσπισης από το βρετανικό πλαίσιο μιας ισχυρής ανεξάρτητης αρχής παρακολούθησης όπως ανέφερε και ο Κλώτη Μωράης προηγουμένως που θα παρεμβαίνει άμεσα όταν υπάρχουν παράπονα από τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα κλείσω με δύο λόγια σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα που προκύπτει μετά από αυτή την συμφωνία που έχει εγκριθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και θα σταλεί προς εσάς προς έγκριση στις 29 Ιανουαρίου. Πέραν των δικαιωμάτων των πολιτών, υπάρχουν πολλά ακόμα ζητήματα ε, για τα οποία θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε. Ιδίω εδώ αναφέρομαι στο πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, που κατοχυρώνει την, και διασφαλίζει την ενιαία αγορά, αλλά αποτρέπει και την ε, διαμόρφωση ενός ε, φυσικού συνόρου μεταξύ των δύο χωρών. Κατά προβλέπονται έλεγχοι για τα εμπορεύματα που θα μπαίνουν ε, και θα εισέρχονται στην Ιρλανδία. Ε, και προσβλέπω σε συνέχιση της συνεργασίας ε, με τις Βρετανικές Αρχές, ώστε όλες οι παλαιότερες διατάξεις που αναφέρονται στην συμφωνία θα τηρηθούν και θα καταστούν λειτουργικές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπαρνιέ. Δίνω τώρα το λόγο στην ε, κυρία Μπενγκιακ για το Συμβούλιο. Κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουμε βεβαίως το ότι θα περάσουμε σε μια νέα φάση της διαδικασία του Brexit, αλλά πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά την ε, διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών, είτε στην μεταβατική περίοδο, αλλά και στη μελλοντική μας σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσεκτική επιτήρηση του πώς θα εφαρμοστεί το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης στο ΕΒ Βασίλειο και στα 27 κράτη-μέλη. Έτσι ώστε οι επιλογές που έκαναν οι πολίτες και οι οικογένειές τους με βάση την ελεύθερη μετακίνηση να προστατευτούν. Άρα βασιζόμαστε στην συνεργασία σας επ' αυτού και σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ψήφισμα από την συζήτηση αυτή. Θα το ψηφίσουμε αύριο. Καλώς απόγευμα.